την έκθεση της κυρίας Φερέρα. Τον λόγο έχει ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο κύριος Βενιζέλος. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα στο πλαίσιο των όσων έχουν συμφωνηθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πριν την ψηφοφορία να κάνω εκ μέρου του Συμβουλίου την ακόλουθη δήλωση. Regarding the ratification of the intergovernmental agreement σε ό,τι αφορά την κύρωση τη διακυβερνητική συμφωνία, θα ήθελα να επιβεβαιώσω εκ μέρου του Συμβουλίου ότι υπογράφοντα τη συμφωνία αυτή για τη μεταφορά και αμοιβοποίηση των συμφορών προ το ενιαίο Ταμείο Εξυγίαση είναι έτοιμοι να δηλώσουν ότι θα προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία κύρωση σύμφωνα με τα αντίστοιχα με τι αντίθυνε εθνικέ του υποχρεώσει και διατάξει, προκειμένου να επιτρέψουν στον ενιαίο μηχανισμό εξυγίαση να είναι πλήρω λειτουργικό από την 1η Ιανουαρίου του 2016. Ευχαριστώ. Το λόγο για ο Επίτροπο Μπαρνιέ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε κάποια λεπτά έτσι ώστε ε, να ε, μπορέσω και εγώ να ευχαριστήσω όπως και εσείς άλλωστε κύριε Πρόεδρε Σούλτς στους ε, βουλευτές που εργάστηκαν επί τη βάση εκθέσεως και των Σκιωδών. Σήμερα το πρωί είχα την ευκαιρία να κάνω μια καλύτερη αξιολόγηση των 41 κειμένων που αφορούν ακριβώς αυτά τα κείμενα στα οποία καταλήξαμε κύριε Πρόεδρε μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και με τη στήριξη βεβαίως διαφόρων Προεδριών και της Ελληνικής Προεδρίας φυσικά. Αυτό αυτό αποτελεί πραγματικά ακρογωνιαίο λίθο για την σταθερότητα ε, της ε, Ευρωζώνης, γιατί η σταθερότητα της Ευρωζώνης ε, σημαίνει σταθερότητα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλάβαμε λοιπόν τις ευθύνες μας και αναλάβαμε και την ευθύνη του να ξαναβάλουμε μια φρασεολογία, ένα λεξιλόγιο το οποίο περιλαμβάνει και την ηθική και τη δεοντολογία ε, ε, λεξιλόγιο που είχαμε ξεχάσει. Εδώ και 30 χρόνια αγωνιζόμαστε για τα θέματα αυτά και τελικά χάρη σε όλους σας ε, καταφέραμε κάτι. Αναφέρθηκα σε 41 κείμενα τα οποία προέρχονται από όλο το φάσμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που όλοι λοιπόν ε, έβαλαν το λιθαράκι τους έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το ε, ρυθμιστικό οικοδόμημα το οποίο θα δώσει σταθερότητα, ε, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ζολή, ζητήσατε το λόγο. Α, όχι, εντάξει, σαφές, μάλιστα. Περνάμε άρα στην ε, ψηφοφορία πρώτα απ' όλα για το συνολικό κείμενο τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η πρόταση της Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε σε ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. ...570 υπερψήφισαν, 88 κατά, 13 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Φερέιρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με τις ψηφοφορίες. Ο κύριος ε, Σιλβέστρη ζήτησε το λόγο. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Πολύ ωραία. Προχωράμε λοιπόν. Έκθεση Βάιντεν Χόλτσερ. Ενιαία ε, ψηφοφορία, διονομαστικής κλήσεως, άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Βόρτμαν Κόλ. Διονομαστικής κλήσεως άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Κορέιρα Κάμπος. διονομαστικής κλήσεως. Άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται. Έκθεση Σπερώνη. Ε, ψηφοφορία διονομαστικής κλήσεως, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Νίτρας. Ψηφοφορία διονομαστικής κλήσεως, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αντρές. Διανομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Γκάλο. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έκθεση Ντερντάν. Διονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ακόμα μια έκθεση Ντερντάν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Σάιμον. Η θέση του Συμβουλίου είναι εγκεκριμένη. Έκθεση Φιντάντσα, πρώτο μπλοκ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πρόταση της Κομισιόν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα διονομαστικής κλήσεως άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Απροβάτο. Εγκρίνεται. Έκθεση Λάιχτφριντ. Μπλοκ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 δέλτα διονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Τροπολογία 72 καταπίπτει, τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 70, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. 10D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 71 καταπίπτει. Ψηφίζουμε την πρόταση της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα διανομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Χέκμαρκ. Μπλοκ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπλοκ 2 καταπίπτει. Πρόταση της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Έκθεση Γκίγκολντ. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα διονομαστικής κλήσεως άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση κλούτε. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η πρόταση της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα διονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Για την έκθεση κλείεται για λογαριασμού πληρωμών η δήλωση της Κομισιόν θα δοθεί γραπτός στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα μπει στα πρακτικά της συνεδρίασης ε, για να την έχετε υπόψη. Επίσης, αν μου επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, δράτω με τις ευκαιρίες να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός πως πολλές δηλώσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγιναν επίσης όσον αφορά την συμφωνία των συνομοθετών για τους εξής φακέλους. Ε, την έκθεση Μπαλτασάρη, για την ε, αποκάλυψη μη οικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών επικοινωνίας από μεγάλους ομίλους ή για την έκθεση Φέρμπερ για τις αγορές ε, χρηματοπιστωτικών ε, μέσων, έκθεση Κέρν για θαλάσσιο εξοπλισμό και για την έκθεση Ροϊτοβα για εξοπλισμό που λειτουργεί υποποίηση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έκθεση Μπερές, μπλοκ 1. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα. Διονομαστική κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Έκθεση Τάιν. Νομοθετικό ψήφισμα διονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεμπάκερ, μπλοκ 1, τροπολογία 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μπλοκ 2, καταπίπτει, πρόταση της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα διονομαστικής κλήσεως άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Χέρτζοκ. Μπλοκ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το μπλοκ 2 καταπίπτει. Πρόταση της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα διονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Βόρτμαν Κόλ, μπλοκ 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το μπλοκ 2 καταπίπτει. Πρόταση της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα διονομαστικής κλήσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Χεράντς Γκαρθία. Μπλοκ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η πρόταση της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα διομοναστικής κλίσεως. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Τούρμες, μπλοκ 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πρόταση της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, νομοθετικό ψήφισμα διανομαστικής κλήσεως. άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Ράνσντορφ, μπλοκ 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα διανομαστικής κλήσεως άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Τζαβέλα, μπλοκ 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα διονομαστικής κλήσεως, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Ford, Μπλοκ 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πρόταση νομοθετικού περιεχομένου η διανομαστικής κλήσεως ε, άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Μπαλντασάρε. Μπλοκ 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση της Κομισιόν. Υπέρ αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα. Διονομαστικής κλήσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση Μπαλντασάρε, μπλοκ 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Ιακολίνο. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρώτο τμήμα ε, σχετικό άρχεται η ψηφοφορία διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επομένως ε, καταπίπτει τροπολογία 6, τροπολογία 2 διονομαστικής κλίσεως, ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 1, το αντίστοιχο τμήμα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3, υπέρ κατά αποχές, απερίφθη ηλεκτρονική υπαλλήθευση για το 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές. Νομίζω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Πρώτο τμήμα ε, της αιτιολογικής σκέψης 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 4 καταπίπτει, επομένως τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Πρόταση της Επιτροπής Διονομαστικής Κλήσεως άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται πρόταση νομοθετικού περιεχομένου, ψήφισμα συγγνώμη, ε, άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση Έλερ, μπλοκ 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 67, διονομαστικής κλίσεως, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 68 διονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Πρόταση της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα διονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Βανίστελόι. Μπλοκ 1. Παρακαλώ. Κυρίες ε, και κύριοι, αυτό το οποίο ψηφίζουμε εδώ πέρα στη δική μου έκθεση και τις ε, υπόλοιπες αφορά τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουμε κάνει ποτέ για την έρευνα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη και το μέλλον στην Ευρώπη πάνω από 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που εργάστηκαν για αυτό το θέμα και για τον ορίζοντα 2020, ιδιαίτερα την Τερέζα Μαδουρέλ, τη συνεισηγήτρια και την κυρία Γκρέσα Καρβάγιο, η οποία επί χρόνια ασχολήθηκε με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Έρευνας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Μπλοκ 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 82, διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 83 διονομαστικής κλήσεως άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Πρόταση της Κομισιόν υπέρ εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα διονομαστικής κλήσεως άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Έκθεση Τόμσεν, μπλοκ 1, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Πρόταση της Επιτροπής, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα, δύο νομαστικής κλήσεως, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ριέρα Μαδουρέλ, μπλοκ 1, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 59 διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 60 διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 61 διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 διονομαστικής κλίσεως άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Ψηφίζουμε την τροπολογία 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 63 διονομαστικής κλίσεως άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 64 διονομαστικής κλίσεως άρχεται. Πέρας. Απερίφθη 65. Διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη 66. Διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη Τροπολογία 67 διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 60, συγγνώμη, 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 69 διονομαστικής κλίσεως άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Πρόταση της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα διονομαστικής κλίσεως άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Ρούμπιχ. Μπλοκ 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα. Δι ονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Παναγιώτοφ, μπλοκ 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, πρόταση της Επιτροπής, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, νομοθετικό ψήφισμα, δύο ονομαστικής κλίσεως, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Γκουαλτιέρη. Τροπολογία 3, υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, μάλιστα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απερίφθη. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 8 διονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απερίφθη. Τροπολογία 2 διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται. Πέρας. Η τροπολογία 2 απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 διονομαστικής κλίσεως άρχεται. Πέρας. Η τροπολογία 9 εγκρίνεται. Τροπολογία 10 διονομαστικής κλίσεως άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 22 υπάρχει μια προφορική τροπολογία του κυρίου Γκουαλτιέρη. Παρακαλώ κύριε Γκουαλτιέρη. Θα ήθελα να καταθέσω αυτή την ε, τελείως τεχνική προφορική τροπολογία. Να προσθεθεί στην παράγραφο 22 το εξής οι οποίοι είναι επιλέξιμοι για καταγραφή και αναμένεται να καταγραφούν για να ευθυγραμμιστεί με τις υπόλοιπε παραγράφου. Ευχαριστώ. Εάν ε, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ε, θα το ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 διονομαστικής κλήσεως άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται απόφαση, ψηφοφορία επί της αποφάσεως, διονομαστικής κλήσεως άρχεται, πέρας. Απροβάτο. Ε. Εγκρίνεται. Έκθεση ΕΡΗ. Τροπολογία 1. Διανομαστικής κλήσεως. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Τροποποίηση 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψήφισμα στο σύνολό του διονομαστικής κλήσεως άρχεται πέρας εγκρίνεται Δεν και Καλφίν τροπολογία 1 διονομαστικής κλήσεως άρχεται η ψηφοφορία πέρας Απερίφθη. Τροπολογία 2 διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Αρχικό κείμενο διονομαστικής κλίσεως. Παράγραφος 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα διονομαστικής κλήσεως άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Αρχικό κείμενο. Χωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα ε, άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 16, ε, πρώτο τμήμα διονομαστικής κλίσεως, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές, ε, εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται αρχικό κείμενο του 22 διονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία πέρας Εγκρίνεται παράγραφος 24 αρχικό κείμενο πρώτο τμήμα διονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 αρχικό κείμενο διονομαστικής κλήσεως άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται 32 αρχικό κείμενο διονομαστικής κλήσεως άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται 35 αρχικό κείμενο διονομαστικής κλήσεως άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται δέλτα αρχικό κείμενο διονομαστικής κλίσεως άρχεται πέρας εγκρίνεται το ψήφισμα διονομαστικής κλίσεως άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια σε όλους τους εισηγητές.